darf sie bitten platz zu nehmen meine damen und herren! καθίστε παρακαλώ κυρίες και κύριοι. Σας ευχαριστώ. Κύριε Πρόεδρε της της Αρχικής Δημοκρατίας σας καλώς ορίζω κύριε Ζέμαν είναι μεγάλη τιμή να σας καλωσορίζουμε εδώ σήμερα αναλάβετε το αξίωμά σας με έναν στόχο τον στόχο να ενισχύσετε την ευρωπαϊκή πορεία της τσεχικής δημοκρατίας και να ξαναφέρετε τη χώρα στο κέντρο της ευρωπαϊκής πολιτικής. Γι' αυτό σας αξίζει μια μεγάλη αναγνώριση και αναμένουμε βεβαίως την ομιλία σας. Έχετε τον λόγο.